della, che, della scuola fatte per eh, ridurre la disoccupazione giovanile hanno sempre in tutti i paesi aumentato la disoccupazione giovanile. Grazie. Vielen herzlichen Dank. Frau Bild, möchten Sie? Oui, euh, moi je pense qu'il faudrait aussi reparler du rôle des parents, parce qu'on a un peu évincé les parents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 konkrétně pracovat. Takže jsem moc ráda, že autorem bude Kristina a těším se na spolupráci. Solo Vielen herzlichen Dank. Poche parole, poche parole per dire intanto grazie a Cristina Ribacca perché mi sembra che la sua impostazione sia un'impostazione assolutamente condivisibile e molto ambiziosa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 dass sie die Antworten und die Anmerkungen der Kolleginnen und Kollegen nur in Englisch äh, übermittelt bekommen. Sie haben jetzt das Wort für fünf Minuten. Herr Schuntes, bitte. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Παρά τις δυσκολίες που εξέθεσε η Πρόεδρος όσο αφορά τα προβλήματα που έχουμε στη διερμηνία, με καλή θέληση και πρόσθετα μέτρα που έχουμε λάβει θα καταφέρουμε να συνονιθούμε. Άρωστε αγαπητοί συνάδελφοι, θεωρώ το θέμα της συγκεκριμένης γνωμοδότησης πολύ σημαντικό για την Επιτροπή μας, όπως είπε και η Πρόεδρος. Τα έργα τέχνης και τα πολιτιστικά αγαθά αποτελούν μέρος της ψυχής και της ταυτότητας ενός λαού, μιας περιοχής, αλλά και αναπόσπαστο κομμάτι της ατομικής και συλλογικής μνήμης και των κοινωνικών και πολιτιστικών αξιών. Γι' αυτό το λόγο σήμερα οι περισσότεροι διεθνείς οργανισμοί και ενώσεις αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στην ε, έννοια της πολιτιστικής... Την τελευταία πρόταση λοιπόν. Γι' αυτό το λόγο σήμερα οι περισσότεροι διεθνείς οργανισμοί και ενώσεις αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στην έννοια της πολιτιστικής κληρονομιάς, στην προστασία, στην ανάδειξη και στη συνέχισή της. Όπως μας έχει δείξει η ιστορία, οι ένοπλες συγκρούσεις και οι πόλεμοι αποτέλεσαν και αποτελούν ορισμένες από τις μεγαλύτερες απειλές για την ακαιρότητα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα έργα τέχνης, οι αρχαιότητες και τα πολιτιστικά αγαθά που λαιλατήθηκαν από νικηφόρους στρατούς αποτέλεσαν λάφυρο και τρόπε πολέμου για τους νικητές ή κατακτητές. Η μεταφορά αυτών των τροπέων στη χώρα των νικητών αποτέλεσε πράξη επισφράγησης της νίκης της υποταγής και της ταπείνωσης του ιτημένου. Στη σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία, αγαπητοί συνάδελφοι, όπως γνωρίζετε, ξεχωρίζει η απεχθής δράση των Ναζί κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και η άνευ προηγουμένου κλοπή, λαιλασία, φαρπαγή και παράνομη διακίνηση έργων τέχνης, αρχαιοτήτων και πολιτιστικών αγαθών που έλαβε χώρα, που συνετελέστηκαν δηλαδή, σε ευρωπαϊκό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Πιο πρόσφατο παράδειγμα πάντα στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο αποτελεί η λαιλασία αρχαιοτήτων από την Κύπρο κατά τη διάρκεια και μετά την τουρκική εισβολή. Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα. Στη χώρα μου, στην Ελλάδα, το συγκεκριμένο αποτελεί, το θέμα δηλαδή αυτό, αποτελεί ένα σημαντικό, σημαντικό και ευαίσθητο θέμα. Καθώς κατά τη διάρκεια πολλών αιώνων, υπογραμμίζω το πολλών αιώνων, όχι μόνο κατά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο αλλά και πολύ πριν έχουν εξαχθεί από την Ελλάδα παράνομα και αθέμητα χιλιάδες εργατέχνε και αρχαιότητε που σήμερα είτε βρίσκονται σε χέρια ιδιωτών είτε σε σημαντικά μουσεία σε ευρωπαϊκές και όχι μόνο πόλεις. Μάρμαρα του Παρθενώνα, Αφροδίτη της Μήλου, Νίκη τη Σαμοθράκης, τα δύο τελευταία γνωστά γάλματα στο Μουσείο του Λούβρου. Τελειώνω λοιπόν την εισαγωγή ευχαριστώντα την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την πρωτοβουλία σύνταξη αυτή τη ε, νομοθετική ε, έκθεση. Τώρα, πιο συγκεκριμένα στη γνωμοδότηση την οποία έχετε μπροστά και με τα όρια που έχουμε όσο αφορά την έκταση της γνωμοδότησης, θέλω να πω ότι επικεντρώνομαι στην πτυχή των μηχανισμών αποκατάστασης και κατ' επέκταση επιστροφής, η οποία είναι η έρευνα προέλευσης των έργων τέχνης και πολιτιστικών αγαθών. Η γνωμοδότηση περιλαμβάνει μια σειρά προτάσει για την ανάλυση πρωτοβουλίων από την Κομισιόν. Το κείμενο ξεκινά υπογραμμίζοντα την ανάγκη συνεχού και ενεργή προώθηση τη έρευνα προέλευση ω εργαλείο για πιο διαφανή και υπεύθυνη αγορά έργων τέχνης και για την αποτροπή λαιλασιών. Στη συνέχεια η γνωμοδότηση προτείνει την εναρμόνιση των κανόνων σχετικά με την έρευνα προέλευση και τη ενσωμάτωση ορισμένων βασικών αρχών της σύμβασης Unitroid του 1995 για τα κλαπέντα ή παρανόμως εξαχθέντα πολιτιστικά αγαθά σε νομοθετική πράξη. Η συγκεκριμένη πρόταση αποσκοπεί στην εξάλληψη του πρόσφορου εδάφους για λαιλασίες και ελαθρεμπορία που δημιουργεί η έλλειψη κοινών προτύπων αλλά και χαλαρή εφαρμογή ή απουσία κανόνων σε ορισμένα κράτη-μέλη. Επίσης με την υιοθέτηση της συγκεκριμένης πρότασης τα κράτη-μέλη οφείλουν να αποδώσουν όλα τα παρανόμως αποκτηθέντα έργα τέχνης που κατέχουν και για τα οποία υπάρχει αίτημα επιστροφής. Ακόμα, η γνωμοδότηση ζητάει τη δημιουργία μιας κεντρικής βάσης δεδομένων που θα περιλαμβάνει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες που έχουν καταστεί ή καθίστανται διαθέσιμες ως συνέπεια της αυξανόμενης έρευνας προέλευσης για την εξακρίβωση του ιστορικού επαναλαμβάνω του ιστορικού κυριότητας των, ενός έργου τέχνης. Λόγω της ευαισθητοποίησης του κοινού για τα λαιλατημένα έργα τέχνης στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και της αύξησης των ετοιμάτων επιστροφής έχουν δημιουργηθεί αρκετές βάσεις ε, δεδομένα με ιστορικά κυριότητας. Με βάση λοιπόν αυτό, συμπυκνώνω λίγο το λόγο μου, με βάση δηλαδή αυτές τις βάσεις δεδομένων που ήδη υπάρχουν, θα πρέπει να εφαρμοστεί ένα κοινό σύστημα καταλαγογράφησης Τέλος, το κείμενο θεωρεί ότι για να διευκολυνθεί η ορθή έρευνα προέλευσης απαιτεί τη δημιουργία ενός εγγράφου ή μητρώου συναλλαγών το οποίο θα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα ονόματα των κυρίων τι χρονικέ περιόδου κυριότητα και μέσα μεταβίβαση. Κατά συνέπεια, ζητάμε από την Επιτροπή να υποστηρίξει αυτέ τι κοινέ κατευθυντήριε γραμμέ σχετικά με τα Μητρώα και να ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη, ούτω ώστε να θεσπίσουν αυτή τη γενική υποχρέωση στους επαγγελματίες της αγοράς. Αγαπητοί συνάδελφοι, τελειώνω. Επικεντρωνόμαστε λοιπόν στη γνωμοδότηση σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα όσο αφορά την έρευνα προέλευσης. Ζητάμε να προωθηθούν αυτοί οι μηχανισμοί αποκατάστασης και χνηλασιμότητας για την αδιαφανή και υπεύθυνη αγορά έργων τέχνης καθώς και για τη διευκόλυνση ετοιμάτων επιστροφής αλλά και η αποτροπή μελλοντικών λαϊλασίων. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Εκτός κειμένου ευχαριστώ τη Φαμπιέν από την Επιτροπή μας που με βοήθησε πολύ ε, ε, σημαντικά για να μπορέσουμε να συντάξουμε και να διαμορφώσουμε αυτή τη γνωμοδότηση. Σα ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ.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 or cultural goods acquisition with the EU is supporting financially any war or conflict. All actors of the market, art market, have a piece of responsibility in preventing it. Thank you. Vielen herzlichen Dank. Frau Bild für zwei Minuten. Donc, je vais essayer de parler doucement et je m'excuse auprès des traducteurs, je suis toujours un peu rapide.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 Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους πήραν το λόγο λέγοντας τις απόψεις τους από ό,τι κατάλαβα ε, συμφωνούν οι σκιώδεις ηγητές με τις βασικές κατευθύνσεις που δίνει η γνωμοδότηση επομένως δεν έχω να κάνω κάποια επιμέρους παρατήρηση ένα σχόλιο ε, ακροτελεύτιο που λέμε τελευταίο ε, επαναλαμβάνοντας, πράγμα που διαπίστωσα και από τις ομιλίες, ότι το θέμα αυτό της προστασίας, πλευρά της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, ακουμπάει στην ψυχή, στον πυρήνα της δουλειάς μας, στον πυρήνα της Επιτροπής μας. Διότι υποθέτω, μάλλον φαντάζομαι και όλοι, ε, ότι η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, εκτός των άλλων, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μιας Ευρώπης των αξιών, θεωρεί υποχρέωσή της, της Επιτροπής μας δηλαδή, να προστατεύσουμε την πολιτιστική κληρονομιά, να παρακολουθήσουμε την ιστορία της εξέλιξης του πολιτισμού. Και είναι πολύ κρίσιμο θέμα και δεν το τονίζω παραπάνω επειδή εγώ είμαι ε, ο εισηγητής, γιατί νομίζω ότι ξαναλέω είναι η καρδιά της, ε, της Επιτροπής μας. Και εδώ η άλλη παρατήρηση είναι αναγκαστικά περιοριζόμαστε στο πώς θα γίνει καλύτερη διαχείριση η προέλευση, η καταγραφή, το ιστορικό μήματος της πολιτιστικής κληρονομιάς. Δηλαδή αυτό που μπορούν να γίνουν εμπορεύματα ή λαιλατούμενα αγαθά ή να το πω με την ορολογία τη δική μας τα αποτελέσματα των οικαστικών τεχνών ζωγραφικής, γλυπτικής που μπορεί να γίνουν εμπόρια. Η προστασία όμως της πολιτιστικής κληρονομιάς αφορά και τις άειλες πλευρές του πολιτισμού. Επομένως η έκκληση είναι να υπερασπιστούμε και αυτή την πολιτιστική κληρονομιά και την πολιτιστική κληρονομιά και των αξιών της Ευρώπης και ένα δείγμα αυτής της ε, προσπάθειάς μας θα είναι αυτό με διορθώσεις και τα λοιπά αλλά να βάλουμε και ένα στίχημα στην Επιτροπή μας να συνεχίσει τέτοιες πρωτοβουλίες για τέτοια θέματα γιατί είναι πάρα πολύ κρίσιμα, είναι ευαίσθητα και συνδέονται και με ε, επίκαιρες εξελίξεις. Και τελειώνω με αυτό, τελειώνω με αυτό ε, το σημείο που ανέφερε ο συνάδελφος, το ανέφερα και εγώ στην εισήγησή μου, είναι γνωστό το ελληνικό παράπονο σχετικά με τα μάρμαρα του Παρθενώνα που εξακολουθούν να φιλοξενούνται στο Βρετανικό Μουσείο στο όνομα ότι δεν υπήρχαν καλά, καλή, καλές προϋποθέσεις να φυλαχθούν στην Αθήνα. Σήμερα δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Αυτά πρέπει να γυρίσουν στην ενότητα και όχι επειδή τα φτιάξαν οι Έλληνες. Εδώ τώρα, σωστά επισήμανε ο συνάδελφος, και γι' αυτό πρέπει να εξοπλιστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με αξίες, θα έχουμε να, τις δυσκολίες ενδεχομένω με τον Brexit. <laughs> Επομένως, δεν το, το κλείνω εκεί για να μην... Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση, να το πω έτσι, θωρακιστεί απέναντι σε τέτοια πράγματα και με τις δυσκολίες του Brexit μπορεί να λυθεί αυτό το πρόβλημα για την υπεράσπιση, ξαναλέω, τη πολιτιστική κληρονομιά, όχι ω μια εμπορική ανταλλαγή, τι δίνει η ΜΕΗ και τι θα δώσουμε εμεί, τι θα πάρουμε από εκεί. Με αυτή την έννοια θεωρώ ότι η δική μα προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί. Σα ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε και για δεύτερη φορά και θα το... η πρόεδρο θα πει τι κάνουμε στη συνέχεια.